να φύγουν αν χρειαστεί. Εγώ δεν το ζήτησα, αλλά σας συγχαίρω και ελπίζω οι άλλοι πρόεδροι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη, δεν ήταν διαδικαστικό αυτό, αλλά επειδή μου φερθήκατε καλά σας άφησα να μιλήσετε. Καλώς. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπή, ο νόμο για τα μέσα ενημέρωση στην Ουγγαρία. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η, Επίτροπη, η Επίτροπος Κρός έχει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, με χαρά μου σας ενημερώνω ότι μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο σήμερα το πρωί στο Στρασβούργο έλαβα τα καλά νέα ότι ο Ούγγρος Πρωθυπουργό συμφώνησε να τροποποιήσει τον νόμο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να συμμορφούνται με όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήσαμε ε, απαντώντας τις ανησυχίες που ετέθησαν όσον αφορά την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ άλλων. Με διαβεβαίωσαν κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ότι οι τροπολογίες θα υιοθετηθούν από την Ουγγρική κυβέρνηση στην επόμενη συνεδρίαση και ε, από ό,τι βλέπω από τους Ούγγρους συναδέλφους ε, σωστά το ανέφερα και θα περάσει και από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο στις επόμενες μέρες. Οι τέσσερις τομείς, ε, κύριε Πρόεδρε, στους οποίους συμφώνησαν ε, να τροποποιήσουν την ομοθεσία τους οι Ούγγροι είναι οι εξή. Πρώτον, ισορροπημένη κάλυψη. Οι τροπολογίες θα περιορίσουν τις απαιτήσει ε, αναφορών ε, για τις μεταδόσεις όπως ε, συμβαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη και δεν θα εφαρμόζονται πλέον αυτές οι απαιτήσει για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες on demand ή στο γραπτό τύπο. Επιπλέον, οποιαδήποτε περιορισμός μετάδοσης θα πρέπει να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εποπτεύει τον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεται η αρχή αυτή σε δευτερεύον δίκαιο, σε δευτερογενές δίκαιο. Αναφέρθηκα σε τέσσερις τομείς. Ο δεύτερος τομέας είναι η αρχή της χώρας ε, καταγωγής. Οι τροπολογίες οι οποίες συμφωνήθηκαν σημαίνουν ότι δεν θα υπάρχει πλέον ε, ε, πρόστιμο για, από, εξω, από τρίτες χώρες ε, για παραβίαση νόμων για την προστασία ανελίκων ή για άλλους λόγους. Οι ουγγρικές αρχές θα μπορούν να αναστείλουν την μετάδοση αυτών των υπηρεσιών στην ουγγρική επικράτεια, κάτι το οποίο συνάδει με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό κύριε Πρόεδρε. Σημαίνει ότι όσοι είναι νόμιμα εγκαταστημένοι και έχουν άδεια σε άλλα κράτη-μέλη και συμμορφούνται προς την ομοθεσία των χωρών αυτών θα μπορούν να μεταδίδουν ελεύθερα στην Ουγγαρία χωρίς να ελοχεύει ο κίνδυνος να ε, τους επιβάλλουν πρόστιμα οι Ουγγρικές αρχές. Τρίτον, καταχώρηση των μέσων. Η τροπολογία σημαίνει ότι ε, η εξωτερική πάροχη ε, μέσω μαζικής ενημέρωσης θα είναι ελεύθερη αφού ε, έχουν περάσει υπηρεσία τους. Αυτό συνάδει με την ε, οδηγία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πρώτερη έγκριση από τις Ουγγρικές Αρχές για να μπορέσει να μεταδώσει κάποιος ένα πρόγραμμα. Τέταρτον, προσβλητικό περιεχόμενο, κύριε Πρόεδρε. Η Ουγγρική κυβέρνηση συμφώνησε να τροποποιήσει και άλλη μία διάταξη του νόμου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δημιούργησε ανησυχίε για την ελευθερία έκφρασης. Υπήρχε μία διάταξη του νόμου που διευκρίνιζε ότι το περιεχόμενο των μέσων δεν θα πρέπει να προσβάλλει εντό εισαγωγικών ακόμα και ε, μέσω υπόνοιας ε, και αναφορά σε συγκεκριμένους ανθρώπους, ε, μειονότητες ή και στον ευρύτερο πληθυσμό. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχει διακριτική συμπεριφορά. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές δεν θα ισχύουν πλέον για όσους παρέχουν προγράμματα μετάδοσης και είναι κατεστημένη σε τρίτες χώρες. Εμείς συνεργαστήκαμε στενά με τις Ουγγλικές Αρχές και θα συνεργαστούμε προκειμένου ε, να υιοθετηθούν οι συμπεφωνημένες αλλαγές και να περάσουν στην εγγλική νομοθεσία και να εφαρμοστούν στην πράξη. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, αλλά αυτό είναι σαφές νομίζω. Και περιττό να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επαληθεύει και τους εθνικούς κανόνες που εφαρμόζουν την οδηγία VMS και σε άλλα κράτη-μέλη και εάν υπάρχουν ανάλογες ανησυχίες ε, θα τεθεί το ζήτημα. Η Κομισιόν, με βουλευτές, δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητες. Δεν φοβάται να ορίσει την ελευθερία των ΜΜΕ και τον πλουρανισμό όπου χρειάζεται. Στην προκειμένη περίπτωση ελπίζω να το αποδείξαμε. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Εκτελεστική Επιτροπή αναγνωρίζει και συμμερίζεται τις ανησυχίες που πολλοί από εσά και τμήματα της κοινωνίας των πολιτών εξέφρασαν όσον αφορά γενικά την κατάσταση των ΜΜΕ στην Ευρώπη και είμαι έτοιμη, Πρόεδρε, να προχωρήσω και να αναλάβω περισσότερη δράση όσον αφορά τον πλουραλισμό των ΜΜΕ μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σεβόμενη την επικουρικότητα. Η Κομισιόν όχι μόνο έχει την υποχρέωση, αλλά ενδιαφέρεται κιόλα να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερόντων και των νομοθετών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μεταβαλλόμενες δομές ε, της το τομέα των ΜΜΕ στην Ευρώπη οδηγεί σε ανησυχίες για το μέλλον γιατί προσφέρει ευκαιρίες αλλά και μεγαλύτερους κινδύνους του πληρορισμού λόγω των, της κατάστασης ιδιοκτησίας. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε να ελέγχουμε τον πληρορισμό των ΜΜΕ σε μευρύ πλαίσιο για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε ε, εντεταγμένα τα μέσα αυτά στο κοινωνικό και οικονομικό τομέα και όχι να τα εξετάζουμε ξεχωριστά. Γι' αυτό, Πρόεδρε, τίνω να οργανώσω μια ομάδα όλων των ενδιαφερομένων για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των ΜΜΕ τώρα και στο μέλλον συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης του πλουραλισμού των ΜΜΕ στην Ευρώπη και ξέρετε ότι πάνω σε αυτό θα ακούσουμε με μεγάλη προσοχή ό,τι έχετε να πείτε. Γι' αυτό θα συμπεριληφθεί, εάν θέλει να δεχθεί την πρόσκληση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα συμμετάσχει στην ομάδα αυτή των εμπειρογνωμών. Τι λεπτομέρειε θα σα δώσω το γρήγορα. Η ομάδα αυτή θα με συμβουλέψει ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά τον τομέα των ΜΜΕ. Και έχω πλήρη δέσμευση να αναλάβω συγκεκριμένε ε, δράσεις μέσα στα πλαίσια όλων των ομαδιτών που έχω. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο. Περνάμε τώρα στους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Πρώτα για το Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Σκούρια για δύο λεπτά. <clears throat> Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είμαι σε δύσκολη θέση ε, για τη συζήτηση αυτή, διότι ουσιαστικά η Επίτροπος μας είπε ότι είναι άχρηστη συζήτηση, διότι δεν υπάρχει πλέον ε, λόγος να αμφισβητούμε κάτι, διότι όπως ε, κατά πάσα πιθανότητα αν μας είχαν ακούσει και άλλοι συνάδελφοι είχαμε πει και επανειλημμένως στη διάρκεια των συνεδριάσεων των Επιτροπών αλλά και εδώ στην Ολομέλεια ίσως θα έπρεπε να περιμένουμε λίγο. Στο κάτω-κάτω της γραφής η Ουγγρική κυβέρνηση ήταν πάντα διατεθειμένη να απαντήσει και να δεχτεί τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήταν περίεργο το αντίθετο για μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή ε, ασκεί και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να μην ακολουθεί λοιπόν τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν μάλλον περίεργο. Παρ' όλα αυτά αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Υπήρχαν ε, κάποια στοιχεία πέραν των ιδεολογικών, υπήρχαν και πολιτικοί λόγοι για τους οποίους έπρεπε να γίνει αυτή η συζήτηση και παρουσιάστηκαν και ψηφίσματα ε, τα οποία ε, θα έπρεπε να ψηφίσουμε αύριο. Ε, ίσως θα έπρεπε να περιμένουμε μάλλον να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στις ε, δημοκρατικά εκλεγμένες ε, κυβερνήσεις από τους λαούς, ε, κυρίως τον Ουγγρικό λαό, ο οποίος έδωσε τόσο μεγάλη πλειοψηφία στην κυβέρνησή του, ένα τόσο μεγάλο ποσοστό που δεν χρειαζόταν να χειραγωγεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας του η Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να ζητήσουμε από του ε, σοσιαλιστέ και φιλελεύθερου συναδέλφων που παρουσίασαν συγκεκριμένα ψηφίσματα να αναστείλουν τα ψηφίσματα, να μην ε, γελιοποιηθούν και να αποσύρουν τα ψηφίσματα, να αφήσουν το Κοινοβούλιο να συνεχίσει τι εργασίε του για πραγματικά προβλήματα τα οποία χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτε. Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο για το έργο τη. Ο κύριος Μωράες για τρία λεπτά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 Πρόεδρε, η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών προφανώς καλωσορίζει την πρόοδο στις τέσσερι βασικούς τομείς ε, δηλαδή την χώρα προέλευση, την καταχώρηση κτλ. Και ε, εξάλλου αυτά έλεγε το δικό μας το ψήφισμα. Ασκούσαμε πίεση σε εσά και στι ε, Ουγγρικές Αρχέ και περιμέναμε αυτά τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω για το χρονοδιάγραμμα. Συγγνώμη, είναι σύμπτωση αυτό που είπατε ότι μόλι περιμένατε εκεί στο αεροδρόμιο, μάθατε τα νέα, ή μήπω η πίεση του Κοινοβουλίου ε, λειτουργήσε γιατί υποβάλαμε τέσσερις βασικές τροπολογίες σε τέσσερις βασικούς ε, τομείς και έτσι κατοχυρώσαμε ε, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ε, γιατί ανάμεσα στην Ουγγρική Κυβέρνηση και στην Επιτροπή. Ε, είναι σαφής η θέση μας ε, και επιβεβαιώνεται, αλλά ε, είναι επίσης σαφές ότι δεν καλύπτονται άλλες βασικές ανησυχίες του Κοινοβουλίου και ειδικότερα της δικής μας της ομάδας. Βασικά ζητήματα εκκρεμούν. η σύνθεση και το χρονοδιάγραμμα για τη συγκρότηση της Επιτροπής ΜΜΕ και νομίζω ότι θα συνεχίσει να ασκείται πολιτική και δικαστική πίεση αν παραμείνει έτσι η σύνθεση αυτής της Επιτροπής. Ε, κατόπιν, ε, λυπούμεθα που δεν ακολουθήσατε τις προτάσεις του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παραβίαση της αρχής της εμπιστευτικότητας ε, για δουλειά των δημοσιογράφων, ε, τις σχετικές κυρώσεις και επίσης την ανεξαρτησία των δημοσίων ειδοσιογραφικών πρακτικών πρακτορείων ε, και καναλιών. Θα θέλαμε απαντήσεις κατά προτίμηση σήμερα. Ε, προφανώς ε, χαιρόμαστε που η Ουγγρική κυβέρνηση ε, κάνει αυτά τα βήματα και ελπίζουμε να εγκρίνει το νομοσχέδιο. Αλλά επίσης ελπίζουμε να καλύψει όλες οι υπόλοιπες ανησυχίες του Κοινοβουλίου σε αυτό το τομέα. Σα υπενθυμίζω και τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ειδικότερα το άρθρο 11 που προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης. Θέλουμε και άλλες απαντήσεις. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι όλα είναι σύνομα, σύμφωνα Λοιπόν το άρθρο 11, ε, η αρχή της διαφάνειας, της ε, λογοδοσίας, οι βέλτιστες πρακτικές ε, πρέπει να κατοχυρωθούν. Έχουμε υποβάλει εμείς το ψήφισμα διότι ζητήσαμε αυτές οι υποχωρήσεις που ήδη επιτύχατε στις διαπραγματεύσεις αλλά όχι μόνο. Θέλουμε ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν πρόκειται να βρούμε δικαιολογίε για κανέναν και θέλουμε να προστατευτούν οι Ούγγροι πολίτες και γενικότερα οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους ε, φιλελεύθερους, η κυρία Βέμπερ για δύο λεπτά. Thank you, Chair. Commissioner... Σας ευχαριστώ Επίτροπε, συνάδελφοι, στο Κοινοβούλιο συζητήσαμε στο, μελετό, στο παρελθόν περιπτώσεις κατά τις οποίες ε, κάποιες κυβερνήσεις έδειξαν την βούλησή τους να ελέγξουν τα ΜΜΕ. Ποτέ δεν είχαν πάει τα πράγματα τόσο μακριά όσο στο νόμο της Ουγγαρίας. Ε, τηλεόραση, ε, ραδιοφωνία, γραπτός τύπος, όλα ελέγχονται, καταγραφή, από δοσή. Τι εκπομπή εμείς ε, στην ομάδα του Ε. είχαμε πρώτη εκφράσει την αντίδρασή μας για το νόμο και μας είχαν κατηγορήσει τότε ότι ήμασταν πολιτικά κινούμενοι αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο γιατί και η ίδια η κυβέρνηση της Ουγγαρίας δέχεται ότι υπάρχουν σφάλματα στο νόμο αυτό και γι' αυτό δέχεται να κάνει πολλές αλλαγές. Ε, πιστεύουμε την Κομισιόν αυτή είναι η αλλαγή της ε, Ουγγρικής κυβέρνησης και ελπίζουμε να τη λάβουμε γραπτά. Ε, Παρ' όλα αυτά, οι τομεί στου οποίου αναφέρθηκε η Κομισιόν είναι ένα τμήμα τη ε, ευρύτερη εικόνα και άλλα ε, τομεί θα πρέπει να αλλάξουν, ιδίω εκείνοι που αφορούν την τεράστια δυνατότητα ελέγχου στα χέρια ενός πολιτικά ορισμένου ατόμου που θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου των ΜΜΕ για εννέα χρόνια έλλειψη προστασίας των πηγών των δημοσιογράφων και λοιπά. Στο κάτω-κάτω όχι μόνο οι επικριτές αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπολογή προς την Ουγγρική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών και τους δημοσιογράφους γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης επέκριναν αυτές τις πτυχές που σας ανέφερα. Δεν μπορούμε όλοι να κινούμεθα από πολιτικά κίνητρα των αντίον κινούμεθα από γενικό συμφέρον να, και ενδιαφέρον να δούμε η ελευθερία των ΜΜΕ να είναι απόλυτη προς όφελος των πολιτών. για λεπτά. Dank u voorzitter. Mijn eerste vragen zijn Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απευθύνω το πρώτο μου ερώτημα προς την κυρία Κρός. Ε, ε κύριε Επίτροπε, η οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα αναφέρει ε, μια ανεξάρτητη αρχή, αμερόληπτη αρχή. Χρειάζεται μια αρχή που να μπορεί να επιβάλλει σημαντικότατες ε, κυρώσεις αν χρειαστεί. Όλα αυτά δε σε, μια εξαιρετικά πολλωμένη, αν θέλετε, ατμόσφαιρα στην ε, Ουγγαρία. Ε, δεν έχει κατοχυρωθεί η ανεξαρτησία αυτής της αρχής. Ε, γιατί δεν Γύρατε αυτό το ζήτημα των αρμοδιοτήτων δηλαδή αυτού του νέου οργάνου και γιατί δεν το συνδέσατε με το αντίστοιχο άρθρο της ε, Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, καταφέρατε η Ουγγρική ε, κυβέρνηση να περάσει τέσσερις αλλαγές για τα λοδαπά ΜΜΕ και τα λοιπά, αλλά δεν κάνατε τίποτα για τα εγχώρια ε, ΜΜΕ. Οπότε θριαμβολογείτε αλλά νομίζω ότι η κατάσταση δεν θα αλλάξει ε, και θα συνεχίσουν οι αυθαίρετες ε, απαγορεύσεις. Ε, νομίζω ότι δεν μπορείτε να δηλώνετε ικανοποιημένοι με τις εξελίξεις. Τώρα θα απευθυνθώ στο συνάδελφο του ΕΛΚ. Είπατε ότι υπήρξε χειραγώγηση, ότι έγιναν σχόλια Ε, ε, για πολιτικές ε, σκοπιμότητες, μιλήσαμε για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργό Όρμπαν φαίνεται να κατάλαβε ότι πρέπει να τροποποιήσει το σχετικό νόμο. Μα μου θυμίζει την εποχή του Στάλιν, δηλαδή εξαφανίζονταν άνθρωποι, κυκλοφορούσαν παραποιημένες φωτογραφίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να γίνει ένας νέος τέτοιος κρατικός μηχανισμός. Κυρία, κυρία Κύριε, κυρία Μωρά έχει μια μπλε κάρτα, θα τη δεχτείτε. Ε, ναι, πρόεδρε. Αν θέλετε να με ακούσετε, βάλτε ακούσικά σα. Κύριε Στρογγετίνη, ξέρουμε τι έκανε η κυβέρνηση Φίντεξ και πολλοί από τους αριστερού και την ομάδα S&D και ο κύριος Κοντβέντιτ χειροκροτούν τώρα και χαίρονται ότι μπορούμε τώρα, μπορούν τώρα να μας κάνουν μαθήματα για τη δημοκρατία. Τι έγινε όμως το 2006. Πού ήταν όλοι αυτοί οι επικριτές. Το αριστερό κόμματα δεν κάναν τίποτα για να μην φτάσουν σε αυτή την κατάσταση σε σχέση με τις διαδηλώσεις. Ε, κυρία Σογεντίνη, 30 δευτερόλεπτα. Uh, δεν πιστεύω ότι δημιουργούν βία τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν καταλαβαίνω ποια σχέση έχει αυτό που συμβαίνει με την ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας πάντως. για ένα λεπτό. ο λόγος είναι μεγάλη αξία το γνωρίζουν όλοι και γι' αυτό θα πρέπει να συζητηθεί η ελευθερία του λόγου. μου φαίνεται όμως ότι η σημερινή συζήτηση δεν είναι καθόλου σοβαρή. αποτελεί πρόσχημα για τους αριστεριστές και το αριστερό περιβάλλον να επιτεθούν στη δεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού της ουγγαρίας. πράγματι στην ευρώπη μπορούμε να σας δείξουμε πολλές χώρες όπου παραβιάζεται η ελευθερία του λόγου. Αρκεί μόνο να αναφερθούμε στην εμπειρία της Πολωνίας. Στην Πολωνία το κυβερνών κόμμα έχει πλειοψηφία σε όλα τα όργανα που ελέγχουν την εξουσία, στο Κοινοβούλιο, στη Γερουσία, στο φορέα που ελέγχει τα οπτικοακουστικά μέσα και τη δημόσια τηλεόραση, καθώς επίσης και τα ηλεκτρονικά μέσα. Και εκεί οι δημοσιογράφοι απολύονται απλώς και μόνο διότι γράφουν κάποιες συντηρητικές απόψεις. Τα συντηρητικά προγράμματα και τα δεξιά προγράμματα ε, διακόπτονται. Πού είναι ο κύριος Σούλς ε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι γίνεται όταν γίνονται τέτοια παραβίαση στην Πολωνία. Έχουν συμβεί αυτά στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λάιτφριντ έχει μπλε κάρτα για σας κύριε Ζιόμπρο. Θα δεχτείτε την ερώτηση. Έχει μπλε κάρτα για σας ο κύριος Λέχτρη. Θα τη δεχτείτε. Παρακαλώ, 30 δευτερόλεπτα. Συνάδελφε, αν κατάλαβα σωστά, είπατε ότι σε πολλές χώρες στην Ευρώπη υπάρχει περιορισμός ε, της ελευθερίας άποψης και ελευθερίας τύπου. Ποιες χώρες έχετε κατά νου και τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε κατά. 30, 30 δευτερόλεπτα κύριε Ζιόμπρο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η ελευθερία του λόγου είναι θεμελιώδες πρόβλημα. Αν αρχίσουμε τη συζήτηση θα πρέπει ε, να δούμε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι εξάρτητο των πολιτικών συμπαθειών. Εάν ένας δημοσιογράφος ε, δεν μπορεί να μιλήσει είτε γιατί έχει αριστερές ή συντηρητικές απόψεις θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Ε, οι δημοσιογράφοι στην Πολωνία σήμερα ε, χάνουν τη θέση τους διότι έχουν συντηρητικές απόψεις. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν Λοιπόν, τι κάνει ο κύριος Σούλτς και οι υπόλοιποι που έχουν πιο αριστερές απόψεις όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι πολιτικό το παιχνίδι. Δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο γι' αυτό. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις όπου και να συμβαίνουν. Ακόμα και αν συμβαίνουν στην Πολωνία. Προ όλου, όταν χτυπώ το σφυράκι μου, σημαίνει ότι τελείωσε ο χρόνο σα. Δεν θα πρέπει να δημιουργείτε σύγχυση. Όταν χτυπώ το σφυράκι μου, ε, τελειώνει ο χρόνο αγόρευσή σα, αλλιώ θα σα κλείνω το μικρόφωνο. Usually Συνήθως στο τέλος της συζήτησης. Επίτροπε, άκουσα με πολύ προσοχή αυτά που είπατε και με σοκάρει αυτό που κάνει η Επιτροπή επίτηδες ε, το έκανε η Επιτροπή να πέσει στην παγίδα της Ουγγρικής κυβέρνησης ή όχι. Τι ζητούν κάποιε λεπτομέρειε, κάποιε μικροϋποχωρήσεις και δεν αλλάζουν ε, το νόμο ε, επί τη ουσία. Ε, ε, είναι δυσανάλογα τα μέτρα. Με αυτή την Επιτροπή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θα αρχίσουν να ασφικτιούν τα ΜΜΕ. Δεν πρόκειται να, να ζημιωθεί καμιά αλλαγή. Είναι ντροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να επιτύχει αυτούς, αυτές τις υποχωρήσεις και όλοι το επικροτούν σε όλες τις εφημερίδες και όλα καλά και όλα ωραία. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να υπάρχει λογοκρισία και να παραβιάζεται η ελευθερία τη έκφραση σε οποιαδήποτε χώρα τη Ένωση. Και τώρα δηλαδή δεν έχουμε να παρακολουθούμε μόνο την Ουγγρική κυβέρνηση αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πραγματικά είναι ντροπή αυτό που, ε, που κάνετε. Ο κύριος για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη σελίδα της κοινοβουλευτική ιστορίας δεν θα πρέπει μάλλον να την έχουμε άρρηκτα συνδεδεμένη στη μνήμη μας. Ε, τα όσα συνέβησαν ε, στην στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάφορη υποτίθεται παραβίαση της Ουγγρικής ε, κυβέρνησης ε, του νόμου των μέσων μαζικής ενημέρωσης τελικώς αποδείχθηκε τι έγινε. Πρόκειται για κάτι το οποίο προέκυψε από μια ιδεολογική προκατάληψη και είναι εξίσου επονίδιστο όταν γίνεται ε, ενώπιον μιας χώρας που έχει ε, στο DNA του εγγεγραμμένο την αίσθηση και την ε, μάχη για την ελευθερία. Θα το θυμόμαστε όλοι. Οι πολιτικές δυνάμεις που προήγαγαν αυτή τη συζήτηση η οποία κανένα λόγο ύπαρξης δεν έχει προσπάθησαν να χειραγωγήσουν μια κατάσταση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο και προέκυψε μια κατάσταση από ιδεολογικούς και μένω λόγους. Ακόμα και το γεγονός ότι επισκιάστηκε σαφής λόγο η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ιστορική σημασία για μια πρώην κομμουνιστική χώρα που σήμερα προχωρεί μαζί μας στη μάχη για την ελευθερία. Πρώτα ο κύριος Μπούσουτιλ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Υπό το φως των αγγέλειας που έκανε η Επιτροπή σήμερα είναι σαφές ότι αυτή η συζήτηση έχει ξεπεραστεί από τα γεγονότα και δεν υπάρχει πια καμία βάση να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία για το ψήφισμα αύριο. Πιστεύω ότι εκεί που εξέφρασαν πραγματικές ανησυχίες για το νόμο των ΜΜΕ δικαιούνται απάντηση. Αυτό που μου φαίνεται όπως ανησυχώ είναι ότι αυτό το σώμα προχωρήσει στα προφορία κατά συγκεκριμένων κρατών μελών. Ε, στην περίπτωση αυτή πρόκειται για μια κυβέρνηση ΕΛΚ και πριν εξετάσει ακριβώς τα πράγματα η Κομισιόν και καταλήξει σε συμπεράσματα. Και όλα αυτά έγιναν παρόλο το γεγονός ότι είχε αναλάβει η γκρική κυβέρνηση σε ανώτατο επίπεδο ότι αν η Κομισιόν έβρισκε κάποια σφάλματα στον νόμο προτίθεται να τον αλλάξει, όπως και γίνεται. Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος της συζήτηση αυτής και ποιο είναι το αντικείμενο του ψηφίσματος αυτού αύριο εκτός από πολιτική χειραγώγηση. Το ΕΛΚ, κύριε Πρόεδρε, παραμένει αυστηρά προσκολλημένο στην δέσμευσή του για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου άσχετα από το εν λόγω κράτος μέλος. Δεν τίθεται θέμα. Από την άλλη μεριά δεν προτίθεται να απομονωθούν συγκεκριμένες χώρε μέλη και να καταδικαστούν σφαιρικά πριν έχει ολοκληρωθεί η σωστή νομική διαδικασία. Και όταν ολοκληρωθεί θα πρέπει να τις διβαστούν. Όταν για πρώτη φορά ετέθη το θέμα το περασμένο μήνα, είπα ότι το να πολιτικοποιήσουμε το θέμα αυτό δεν ήταν επίθεση κατά ενό κράτου μέλους, αλλά υπέσκαπτε και την ε, κοινοτική προεδρία. Τώρα υποσκάπτουν νομίζω και το δικό μα ε, θεσμικό όργανο και αυτό δεν επιτρέπεται. Κάνω έντονη έκκληση σε όλε τι πολιτικέ ομάδε να αποσύρουν τα ψηφίσματα που έχουν υποβάλει προς πληροφορία για αύριο, να τι αποσύρουν, όχι να τι αναβάλουν γιατί δεν υπάρχει πια βάση για την ψηφοφορία αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για δύο λεπτά η κυρία Μπαντία. Κύριε Επίτροπε, εκπρόσωποι του Συμβουλίου, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια επανάληψη, αλλά ορισμένε φορέ είναι ε, σημαντικό να επαναλαμβάνονται αυτά τα πράγματα. Η ελεύθερη κυκλοφορία νέων και ειδήσεων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ σήμερα. Αν είναι η ησυχία που εξέφρασε ε, ο ΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ήταν τόσο επίμονε, ήταν γιατί διακυβεύονταν και διακυβεύονται ακόμα ρίζες του ευρωπαϊκού προγράμματος. Εμείς θεωρήσαμε ότι η Ουγγρική νομοθεσία η οποία ε, νεκρήθη κατεπηγόντως από την Ουγγρική κυβέρνηση δεν ε, είχε εξεταστεί καταλήλως και έπρεπε να τροποποιηθεί για να προσαρμοστεί και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και στο βασικό πνεύμα το οποίο εκφράζεται από τις συνθήκες. Ευχαριστούμε και είμαστε ικανοποιημένοι που διαπιστώνουμε και ακούμε σήμερα την Επίτροπο ότι η Ουγγρική κυβέρνηση είναι διατεστημένη να τροποποιήσει την νομοθεσία, αλλά η δημιουργία μιας αρχής ελέγχου των πληροφοριών ε, και ε, ο έλεγχος ενός συμβουλίου όπως θα γίνεται μόνο από μέλη της ε, κυβέρνησης μπορεί να δημιουργήσει ένα πολιτικό έλεγχο που θα οδηγήσει στη λογοκρισία και σε κάτι το οποίο είναι ακόμα χειρότερο στην αυτολογοκρισία. Θα αλλάξετε λοιπόν αυτή τη διάταξη, θα αλλάξει αυτή η διάταξη. Μαζί με την Επίτροπο ε, μοιραστήκαμε τις ανησυχίες μας για την ε, ε, πολυφωνία της ενημέρωσης, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας έκφρασης και των ενημέρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 11 της Χάρτατος των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αλλά οι απαντήσεις που μας έδωσε η Ουγγρική κυβέρνηση, η οποία δέχτηκε να τροποποιήσει το νόμο, θα πρέπει να ελεγχθούν καταλήλως ώστε να φροντίσουμε να αλλάξουν εις βάθος και να μην υπάρχει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα αυτό που σας είπα μόλις για την αρχή ελέγχου. Ε, απαιτούμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις ερευνές της, κυρίως για τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ζητώ συγγνώμη τους από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και από την Επίτροπο, αλλά το θέμα αυτό δεν είναι πολιτικό όπως προσπαθούν κάποιοι να το παρουσιάσουν, αλλά είναι θέμα προάσπασης των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σεβασμού των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην έχετε καμία αμφιβολία, γι' αυτό δεσμευόμαστε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, είναι λίγο παράξενο που ε, ως ε, φιλελεύθερος θα κάνω τη δήλωση που θα κάνω. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν συμφωνώ με την ελευθεροτυπία. Κοιτάξτε, όπως είδαμε και από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων του ΕΛΚΑ, πρόκειται για ένα πολιτικό ζήτημα. Ε, θα ήθελα να ξέρω ε, ποια είναι η απάντηση της Ουγγαρίας ε, στα ερωτήματα που της έχουν τεθεί. Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης. Πάντοτε αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις, αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτήν τη νέα επιτροπή για τα ΜΜΕ στην Ουγγαρία. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει τη σωστή λύση, γιατί δεν επαρκεί μόνο να έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή. Μπορείτε να εμβαθύνετε σε αυτό το ζήτημα. Ε, ένα λεπτάκι, λέει ο Πρόεδρο, για όσου δεν γνωρίζουν τη διαδικασία, είναι, επαφείται στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου το αν θα χωρίσω χώρο, χρόνο για ένα ερώτημα βάσει τη ε, μπλε κάρτα. Ε, αν κρίνω ότι έχουμε χρόνο, το κάνω. Οπότε δεν μπορώ πάντοτε να σα δίνω το λόγο. Ε, ε, επαφείται, ξαναλέω, στη δική μου διακριτική ευχαίρεια και τη διακριτική ευχαίρεια τη γραμματεία. Κυρία Τρούπελ. Κυρίε και κύριοι, δεν υπάρχει κανένα ε, λόγο να αισθάνεται το ΕΛΚ τέτοια ικανοποίηση. Το υπάρχει, έχουν τώρα αλλαγέ στην Ουγγρική νομοθεσία, δικαιώνει εκείνε που το ζήτησαν. Ο κύριο Ορμπαν δεν ήταν από εκείνου που το ήθελαν εκ μια αρχή. Το λέω ξεκάθαρα ότι οι αλλαγέ που υπάρχουν τώρα δεν είναι επαρκεί ή ακόμα έχουμε μία ε, ομάδα, μία αρχή εποπτείας για εννέα χρόνια που θα συμμετάσχουν αυτοί μόνο μέλη του ΦΙΝΤΕΣ. Δεν πρόκειται λοιπόν για δημοκρατική διαδικασία. Κυρία Κρούς, κατά τη γνώμη μου, δεν ε, φτάσατε εκεί όσο μακριά έπρεπε γιατί εσείς ενδιαφερόστε να υπάρχει ησυχία και να μην παρεμποδιστεί η Ουγγρική Προεδρία και όχι τόσο να υπάρχει μια καλή νομοθεσία ΜΜΕ. Θα ήθελα να σας υπέθουμε τον Σοκόντα Μεσέλα, Μιχαήλ Βόντα, που είχαν ζητήσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να τους υποστηρίξουν. Ακόμα δεν το κάνουμε. Αυτή η νομοθεσία κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τύχει νέας δημοκρατικής επεξεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι η Ουγγρική κυβέρνηση στο θέμα αυτό απέδειξε ότι είχε μεγάλη ευαισθησία ενώπιον της Ευρώπης και των αρχών που τη θεμελιώνουν. Πράγματι, αμέσω μετά την έγκριση του νόμου για τα μέσα μαζική ενημέρωση τη Ουγγαρία, ξεκίνησε μία εκστρατεία από τι αριστερέ παρατάξει που χρησιμοποίησε ε, τον όρο όμο, ε, νόμος ε, λογοκρισίας. Μόνο όσοι γνώρισαν το φασισμό γνωρίζουν τι είναι ο νόμος λογοκρισίας. Ενώ οι δημοκρατικές κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι η ελευθερία και η πολυφωνία της ενημέρωσης οικοδομούνται από τη δημοκρατία αλλά θα πρέπει να εναρμονίζονται με όλες, όλες τις εξουσίες ε, του κράτους δικαίου και δεν θα πρέπει να παραβιάζεται το θελμέλιο της δημοκρατίας που είναι η ανθρώπινη ζωή. Το Σύνταγμα της Ιταλίας, το άρθρο 21, διασφαλίζει την ελευθερία ενημέρωσης αλλά απαγορεύει απευθείας και την ε, ε, διαφήμιση. Πρόκειται για ένα νόμο ε, τη διαφήμιση κατά της ζωής των ανθρώπων. Υπάρχει υποχρέωση στη νομοθεσία της Ιταλίας, όχι της πρόερης καταχώρησης, αλλά ε, μια αντίστοιχη καταχώρηση με αυτή που κάνει ο Ουγγρικός νόμος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαίως διατύπωσε ανησυχίες και αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από το συγκεκριμένο δεδηλωμένο στόχο της νομοθεσίας της Ουγγαρίας. Και ο σεβασμός είναι ε, σαφής. Η Ουγγρική κυβέρνηση αμέσως δέχθηκε τις επικρίσεις και ανέλαβε την ευθύνη να αλλάξει τον νόμο βάσει των υποδείξεων που τη έγιναν. Ακόμα και η δήλωση ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εγγραφούν στο Ουγγρικό Σύνταγμα αποτελεί απόδειξη της ε, βούλησης της Ουγγαρίας να ενταχθεί στην ε, ευρωπαϊκή κουλτούρα. Επομένως δεν καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζεται πλέον αυτή η συζήτηση. Γίνεται μόνο για να αναγνωρίσουμε ε, την ευθύνη της Ουγγαρίας που δήλωσε δημοκρατικά ε, έλαβε μια πλειοψηφία η Ουγγρική κυβέρνηση των δύο τρίτων του λαού ε, και επομένως αυτό δεν θεωρώ ότι πρόκειται για λόγο για τον οποίο θα πρέπει να του επικρίνουμε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ την Ουγγρική κυβέρνηση. <clears throat> Ευχαριστώ. Επίτροπε, Υπουργέ, η έκθεση περιορισμού της ελευθερίας των ΜΜΕ είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στην Ευρώπη. Ε, λυπούμε, αλλά ε, έχουν υπάρξει διάφορα τέτοια επεισόδια και έχουν τροφοδοτήσει την ε, συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα. Κοιτάξτε, θα πρέπει να πιέσουμε την κυβέρνηση του ε, Όρμπαν ε, το Σεπτέμβριο. Μας είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο να τροποποιήσουν τη σχετική νομοθεσία τώρα όμως. Υποχρεώθηκαν γιατί έγινε σκάνδαλο αυτή η ιστορία στην Ευρώπη. Τα, οι οικοί κανόνες ε, δεν συνάδουν ε, ε, με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οδηγία για το οπτικοακουστικό υλικό, αντιβαίνουν στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ιτήθηκε η δεξιά κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Πριν από λίγους μήνες είχε κατατεθεί ψήφισμα από διάφορες πολιτικές ομάδες, τα ίδια ισχύουν ως επιτοπλίστων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση. Ε, Πώ θα επηρεαστεί η ελευθερία έκφραση και η ελευθεροτυπία στην Ουγγαρία με τι ε, ε τροποποιήσει ε, του σχετικού νόμου. Γιατί η κυβέρνηση Όρμπαν αποφάσισε να στείλει την ισχύ ε, της τη διάταξη του προηγουμένου νόμου, δηλαδή ότι οι αρχέ πρέπει, η σύνθεση των αρχών θα πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμη εκπροσώπηση όλων ε, των μερών. Τι πιστεύει κυρία Κρός ε, γι' αυτό, γιατί έγινε αυτό επίσης. Ε, δεν θέλω να δημιουργείται αυτή η εθνικιστική ψευδέστηση ότι καταφέραμε να αλλάξουμε την Ουγγαρία. Μην μπερδεύουμε την Ουγγαρία με την Ουγγρική κυβέρνηση και ας μην προσπαθούμε να βάλουμε κάτω από το χαλί το, το, το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν έγινα κατανοητός. Δεν δέχομαι άλλες ε, μπλε κάρτες ε, σε αυτήν την συζήτηση. Ο κύριος Deutsch για δύο λεπτά. Ε, Επίτροπε, στην αρχή της ε, συζήτησής μας είπατε ότι υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στην Ουγγρική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η Ουγγρική νομοθεσία θα τροποποιηθεί σε διάφορα σημεία, αλλά συμφωνώ με τους συναδέλφους μου, ε, η πολιτική αυτή συζήτηση στερείται στόχου και νοήματος. Είναι μια πολιτική πρωτοβουλία της αριστεράς των φιλελευθέρων, την ένα είδος μένους, αυτό διαπιστώ ε, στην αίθουσα σήμερα. Κάποιο από, από την ομάδα των σοσιαλιστών είπε ότι πρέπει να υπεραμεθούμε κάποιων αξιών. Ε, κοιτάξτε, ε, ο Λάρι Φάρη από τους Ούγκρους Σοσιαλιστές ε, είπε ότι είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Ε, ε, και αφήστε που έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. άλλα εφαρμόζονται για τους κομμουνιστές, για τους σοσιαλιστές του Κοινοβουλίου και άλλα για τους υπόλοιπους. κοιτάξτε στο παρελθόν είχαμε διαζητήματα με την σοσιαλιστή η Ουγγρική κυβέρνηση ένας υπουργός αποφάθησε να χρησιμοποιήσει ένα βοηθό του για να εκδώσει οδηγίες προς ένα δημοσιογράφο ε, τελικά παράνομα ε, κατηγορήθηκε για κατοχή ναρκωτικών ο δημοσιογράφος και γίνει σκάνδαλο ε, τότε η Ουγγρική κυβέρνηση αποφάσισε να διώξει ένα δημοσιογράφο για ένα άλλο άρθρο που ήταν επικριτικό ενώπιον της ε, κυβέρνησης. Ούτε τότε ε, ε, είπαμε τίποτα. Επίσης, Ούγγροι δημοσιογράφοι είχαν διερευνήσει κάποια επεισόδια, κάποια, κάποιες απάτες που διαπιστώθηκαν στο Κογκρέσο του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ουγγαρία. Τίποτα δεν είπατε τότε. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί σιωπούσατε και γιατί σήμερα φωνασκείτε ενώ τότε σιωπούσατε. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ καλό που η ευρωπαϊκή κυβέρνηση αποσύρει τα, α, αρνητικά σημεία του νόμου, του νόμου και που εσείς κυρία Κρούση είσαστε εγγνωμένοι αλλά ακριβώ μία μέρα πριν υιοθετηθεί το ψήφισμα για το νόμο ΜΜΕ στην Ουγγαρία είμαστε αναγκασμένοι να βασιστούμε μόνο στη δική σας αξιολόγηση, στην δική σας δήλωση χωρίς να έχουμε τίποτα γραπτό. Εσείς πώς μπορέσετε να καταλήξετε συμπεράσματα αυτά μέσα σε λίγες ώρες. Και ήταν κάποιοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που συνεργάστηκαν εδώ. Γιατί και η όρια αντίδραση της κυβέρνησης είναι ότι αυτές οι αλλαγές δεν θα είναι ουσιαστικέ, αλλά κοσμητικές μορφής. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί σήμερα που συζητάμε το θέμα αυτό, ακούμε ότι θα δράσει η κυβέρνηση σε δύο εβδομάδες και ικανοποιεί αυτό την Κομισιόν. Έχω την εντύπωση ότι Υπάρχουν δικαίω ανησυχίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι οι τεχνικέ αλλαγέ που ανήκει η Ουγγρική κυβέρνηση δεν θα είναι σύμφωνε με τι δημοκρατικέ αναγκαίε αλλαγέ σύμφωνα με τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ανησυχούμε ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, σύνθεση και τις αρμοδιότητες του ελεκτικού σώματος γιατί αυτό θα λέγει τον δημοσιογραφικό έργο. Χαίρομαι που είναι πρόθυμοι να έχουν σε διάλογο μαζί μας, αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν είναι θέμα μόνο της Ουγγαρίας. Εγώ είμαι τέλος δημοσιογράφος. Αυτό είναι για να προστατευτούν όλοι οι δημοσιογράφοι. Η κυρία Ρέντινγκ δεν είναι αρμόδια για αυτό. είναι αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, και θα ήθελα να ξέρω, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το όραμα τη Εκτελεστική Επιτροπή όσον αφορά τη δημοσιογραφία στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ελάχιστα κριτήρια που θα εγγυηθούν την ελευθερία των ΜΜΕ και τον πλουραλισμό η ποιότητα της δημοσιογραφίας ήδη πλήθεται και αλλού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριος Μπέλετ για 1,5 λεπτό. Ε, uh, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, όλοι θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό που η Ουγγρική κυβέρνηση σήμερα διασκεδάζει όλες τις ε, αμφιβολίες που υπάρχουν. Θα υπάρχει ελεύθερος τύπος με πλουραλισμό επίσημη δηλαδή υπόσχεση προς την Κομισιόν θα προσαρμοστεί το δίκαιο αυτό. Ε, όλα αυτά πολύ ωραία είναι, αλλά είναι λυπηρό που μια συζήτηση για τον προορισμό του ΜΜΕ στο σώμα γίνεται πάντα προς την κατεύθυνση ε, εθνικών ε, κομμάτων και κάποιων παιδιών που παίζονται στις εν λόγω χώρες. Είναι πάρα πολύ καλή η πρωτοβουλία αυτή για τον πλουραλισμό στην οποία αναφέρθηκε και η Επίτροπος. Είναι πολύ καλή αυτή η ευκαιρία να καταλήξουμε στη ε, οριστική λύση, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τον πλουραλισμό των ΜΜΕ ανεξάρτητα από οποιασδήποτε εθνικές ε, ανησυχίες. Θα πρέπει αντικειμενικά να δημιουργήσουμε έναν πλουραλισμό, να τον εξετάσουμε εις βάθος. Και θα ήθελα να πω μια πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τον διακανονισμό των ΜΜΕ, όπω είπαν ορισμένοι και όπω αναφέρεται και στο ψήφισμα, δεν θα ήταν η σωστή άγουσα. Ελπίζω να συμφωνείτε, κυρία Προεπίτροπε. Ευχαριστώ. Και εγώ χαιρετίζω την απόφαση της Ουγγρικής Κυβέρνησης να τροποποιήσει το νόμο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η επίθεση κατά της Ουγγαρίας, κατά την άποψή μου, ε, ήταν αβάσιμη και δεν ήταν δίκαιη για την Ουγγαρία. Νομίζω ότι εμείς στην Ευρώπη ορισμένες φορές δεν καταλαβαίνουμε τα πράγματα σαφώς. Ε, η διαδικασία στην Ευρώπη πολλές φορές ήταν ασαφής, ε, η αριστερά ήταν κυρίως επικεφαλής και γι' αυτό υπήρχε το αίτημα για ε, υπάρχει μάλλον το αίτημα για μια πιο ισορροπημένη μετάβαση στις ε, ε, κοινωνίες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία μεταρρύθμισης. Ορισμένοι είπαν ότι η αρχή ελέγχου το μέσο μαζικής ενημέρωσης ε, δεν είναι καλή ιδέα. Αλλά η κυβέρνηση έχει εκλεγεί με πλειοψηφία δύο τρίτων. Ε, έχει δύο τρίτα πλειοψηφία στο, ε, στο Κοινοβούλιο και ορισμένοι δεν γνωρίζουν τους μηχανισμούς για τους οποίους διαμαρτύρονται. η Ουγγρική κυβέρνηση θα φροντίσει τα θέματα των μέσων μαζική ενημέρωσης. Νομίζω ότι εσείς κύριε Επίτροπε θα πρέπει να κάνετε πολύ περισσότερα. Δεν θα πρέπει να κάνετε μόνο τον έλεγχο, αλλά θα πρέπει να κάνετε και ει βάθο ανάλυση σε όλα τα θέματα και αυτό ισχύει και για τη Σλοβενία eye, στα πλαίσια τη διαδικασία Eye θέλετε να θέσετε ένα ερώτημα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά σα είπα ήδη. Σε αυτή τη συζήτηση δεν θα δεχτώ άλλε μπλε κάρτε. Ε, κυρία Φερχέιεν, διαδικαστικό θέλετε λοιπόν. Πολύ ωραία, ένα λεπτό, ορίστε. Πρόεδρε, ε, θέλω να σας ε, θέσω ένα ερώτημα. Ανεξάρτητα από από αυτά που λέτε θα αγωνιστώ για το δικαίωμά σας ε, να τα λέτε, έτσι είπε ο Βολτέρος. Οπότε δεν καταλαβαίνω. Προβλέπεται η παρέμβαση με την ε, μπλε ε, κάρτα και νομίζω ότι δεν ισχύουν τα ίδια για όλους ε, και η δεξιά και η κεντροδεξιά θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να θέσει ερωτήματα όπως έκανε και η συνάδελφη από τα, τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ε, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, αλλά δεν έχει σχέση με την πολιτική ομάδα. Με σειρά προτεραιότητα ε, ε, ε, έδωσα χρόνο στους πρώτους όσοι εκδηλώθηκαν πρώτα. Δεν έχει σημασία η πολιτική ομάδα. Ε, έχουμε και παρεμβάσεις του ενός λεπτού, ελπίζω να τα προλάβουμε όλα και ελπίζω να είχα και το χρόνο τώρα να σας αφήσω να θέσετε το ερώτημά σας, αλλά σας διαβεβαιώ ότι ε, ουδεμία σχέση ε, έχει με κάποια πολιτική επιλογή, αν θέλετε, η απόφασή μου. Η κυρία Φερχέιεν για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, εξαιρετική κυρία Επιτροπή Κρούς, εξαιρετική εκπρόβουση του Συμβουλίου, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω κύριε Κρούς ότι τόσο γλίγορα προωθήσετε την ε, συζήτηση και περάσει διαπραγματεύσει με την Ουγγρική κυβέρνηση. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω την Ουγγρική κυβέρνηση που τήρησε αυτό που είπε σε όλες τις ακρόσεις και συζητήσεις και στην αρχή της ε, συζήτησης. Είπε ότι δηλαδή αν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές θα τις κάνει. Η ελευθερία των ΜΜΕ και ο πλουρισμό των ΜΜΕ είναι οι βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ΜΜΕ έχουν όμω και ιδιαίτερη ευθύνη στην κοινωνία. Θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών, να μην ε, ασκούν διακρίσει και να παρουσιάζουν και την αλήθεια. Δεν κινούνται σε ένα χώρο κενό δικαίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ΜΜΕ έχουν ειδική προστασία, ιδίω λόγω του ε, νομοθετικού πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Κομισιόν νομίζω έχει κάνει πολύ καλά το έργο της ως θεματοπιλακός των ε, συνθήκων εδώ και αν είχαμε περισσότερη εμπιστοσύνη στην εργασία της Κομισιόν δεν θα χρειαζόταν να γίνει αυτή η συζήτηση εδώ σήμερα γιατί το ότι το σύστημα λειτουργεί αποδεικνύει τα αποτελέσματα που μας ανακοινώθηκαν σήμερα ότι θα γίνουν δηλαδή αλλαγές εκεί που το νομοθέτημα δεν ήταν απόλυτα σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οι ιδεολογικέ συζητήσει που συνεχώ ε, διαφαίνονται εδώ, ιδίω σε αυτό το πλαίσιο, είναι περιττέ κατά τη γνώμη μου. Καταδεικνύουν περισσότερο ότι η σωστή ε, εξέταση των επιμάχων σημείων βάσει του ισχύοντο δικαίου μπορούν να διευκρινιστούν με τις απαραίτητες συζητήσεις και τα και ελπίζω οι διάφορες πολιτικές ομάδες να σταματήσουν να παίζουν αυτά τα παιχνιδάκια που παίζουν και να αποσύρουν τα εν λόγω ψηφίσματα. Για λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Η Ουγγρική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία για την τροποποίηση της νομοθεσίας με συγκεκριμένο κείμενο εξ όσων κατάλαβα αλλά επιμένουμε ακόμα να κάνουμε αυτή την ε, άχρηστη συζήτηση. Στην πράξη πρόκειται για μια πολιτική επίθεση σε αυτό το νόμο των ε, μέσων. Στο ψήφισμά σας ζητείτε, ζητάτε σεβασμό ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ και στην ενημέρωση, ενώ η πληροφορίες που διαδίδετε εσείς είναι αβάσιμες, ε, δεν υπάρχει καμία θεμελίωσή τους και το διαπιστώσαμε ακόμα και εδώ στην αίθουσα. Αυτό που ζητάμε είναι δικαίωμα στη μη χειραγωγημένη ενημέρωση και εσείς σήμερα το απόγευμα αυτό το δικαίωμα το έχετε παραβιάσει. Και ε, εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διαπίστωση. Προασπίζεστε αυτή την ελευθερία μόνο όταν μπορείτε να επιτεθείτε στις κυβερνήσεις της δεξιάς μέσω αυτής της ε, ελευθερίας. Αλλά ε, κανείς δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό όταν τον Οκτώβριο του 2006 η σοσιαλιστική κυβέρνηση στους δρόμους της Βουδαπέστης ε, κατά Ε, παραβίασε αυτές τις ελευθερίες ενώ στο νόμο για την ε, χρήση της γλώσσας στη Σλοβακία παραβιάζονταν οι, ε, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Αυτά κατα, κατ' σκανδαλώδη. Αναφερθήκατε σε δικτατορία και σε σχέση με αυτή την νομοθεσία. Εγώ που από μικρή έζησα και την δικτατορία του Τσαουσέσκου ε, έχω την απόδειξη σήμερα ότι για σας η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι μονόδρομος και μάλιστα πολύ συγκεκριμένος. Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ανησυχία μου ε, για την διεξαγωγή της συζήτηση σήμερα. Όλοι ξέρουμε ότι έγιναν παρανοήσεις σχετικά με το νόμο αυτό ε, της Ουγγαρίας. Μα είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκείνη πρέπει να διαλευκάνει την ε, υπόθεση δεν ε, κρίνω σκόπι μια τέτοια συζήτηση στο Κοινοβούλιο, ενώ γνωρίζουμε ότι κάλλιστα μπορεί να βρεθεί λύση τις επόμενες ε, ημέρες. Ε, πρόκειται για μια ιστερική καμπάνια της αριστεράς και πριν από λίγες μέρες δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ αυτό το θέμα. Οι πολιτικοί μας ε, αντίπαλοι χρησιμοποιούν αυτά τα προσχήματα για να επιτεθούν ε, σε μια χώρα όπου πριν από λίγες μέρες ε, κατήγαγε σε ερωτική νίκη συγγνώμη, η κεντροδεξιά. Οι προοδευτικές αυτές δημοκρατικές δυνάμεις εισαγωγικά γιατί σιωπούσαν το 88 όταν στη Σλοβακία η τότε δεξιά κυβέρνηση σε ένα νομοσχέδιο με βαρύτατες ε, ε, κυρώσεις. Ε, λυπούμε ε, και πραγματικά ε, έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά εδώ θα πρέπει να αφήσουμε αυτό το θέμα στα χέρια των ειδικών. Δηλαδή στην Επιτροπή και στην Ουγγρική Κυβέρνηση. Τέλος, θέλω να σας πω το εξή. Το να ε, γίνονται απανοτές επιθέσεις στον Πρωθυπουργό αυτής της χώρας μεσούσης της κρίσης, αυτό μπορεί να πλήξει το εθνικό γόητρο. Προσοχή. Κύριος Καβαντά για ένα λεπτό. Είναι τόσο σοβαρό ε, το θέμα, Πρόεδρε, που πρέπει να υπερβούμε αυτές τις ε, ε, διενέξεις που ακούμε σήμερα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. κοιτάξτε, αγαπούμε την Ουγγαρία και... Θα ήθελαν κάποιοι η διαχείριση των πληροφοριών να γίνεται με πιο ε, δίκαιο τρόπο. Δίκαιο έχουν, αλλά δεν διορθώνουμε την προπαγάνδα με άλλη προπαγάνδα. Α είμαστε σε εγρήγορση λοιπόν. Χαίρομαι που βλέπω ότι πολλά ε, βασικά σημεία ε, θα αναθεωρηθούν, αυτό δέχτηκε η κυβέρνησή σας και θα αναθεωρηθεί ο νόμος το 2001 για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολύ σωστή κίνηση. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε... Ε, ε, χρειάζεται ο σεβασμός ε, της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, μα, αυτό αναζητούσαν οι Ουγγροί στο παρελθόν. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά στα χέρια των ειδικών, στα χέρια της Επιτροπής. Αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, όπως σας είπα, γιατί δεν έχουν επιληθεί όλα αυτά τα ζητήματα. Αφήστε που υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμίσουμε επίσης. Να σας υπενθυμίσω ότι είστε η πατρίδα του Κωσίου του Ζολμπράντα, του Ήρωα του 1940, του Κοπάτσι, του του Σάντορ μαράι, ε, του Ήμερ Κερτές. Ε, μην μας απογοητεύσετε λοιπόν. Ε, μην ξεχνάτε και τον κύβο του Ρούμπικ. Ε, εσείς τον ε, φίβρατε και μην παίζετε με, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως παίζει κανείς με τον κύβο του Ρούμπικ. Ευχαριστώ. Περάσουμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Δυστυχώ δεν θα μιλήσουν όλοι. Να σα αναφέρω τα ονόματα των ομιλητών κατά σειρά προτεραιότητα. Πότε σήκωσαν το χέρι του και κατά πόσον είχαν μιλήσει προηγουμένω. Mr. Galler, Mr. Mauro, Mr. Bostinaru, Mrs. Alfano, Mr. Pasca and Mr. Bronze. There are seven other colleagues that cannot take the floor. I apologize to all of you. Οι δεν θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο. Ζητώ συγγνώμη. Πρώτα ο κύριος Γκάλερ για ένα λεπτό θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός με το χρόνο. Κύριε Γκάλερ, ένα λεπτό. Πού είναι ο κύριος Γκάλερ, έφυγε. Μάικολ Γκάλερ. Δεν ήθελε να μιλήσει. Ωραία. Θα μιλήσει η κυρία Γκαλπέλς για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε. Υπάρχει αυτή η συμφωνία τώρα μεταξύ της Ουγγρικής Κυβέρνησης και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ε, πραγματικά πολύ σάλος έγινε για αυτό τον νόμο για τα ΜΜΕ. Τώρα έχουμε την υπόσχεση προς την Κομισιόν ότι θα υπάρχει αλλαγή. Αυτή η συμφωνία μεταξύ Κομισιών και Εγκορική Κυβέρνηση ισχύει. Καταδεικνύει ότι τα πράγματα βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Ο λόγο για τη συζήτηση αυτή δεν υπάρχει λοιπόν πια. Πολλά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι δεν έχουν πια αντικρίσμα. Δεν δικαιολογείται αυτή η επίκριση. Ορισμένοι αναφέρθηκαν σε σκάνδαλο εγώ νομίζω ότι διεπίτες εκμεταλλεύτηκαν αυτό το θέμα γιατί αυτή η νομοθεσία για τα ΜΜΕ είναι σύμφωνη με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και με όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα πραγματικά να δεχτούμε το θετικό ε, πέρας αυτής της υπόθεσης. Ο κ. Μάουρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακόμα και αν θέλουμε να πιστέψουμε ότι όσοι επέκριναν τόσο στεναρά τον νόμο της Ουγγαρίας θέλουν αποκλειστικό και μόνον ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, νομίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τα όσα έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, από τα όσα ε, συζητήθηκαν στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ε, για την αποφυγή μιας ε, μαύρης σελίδας στο κοινοβουλίο μας και να μην ψηφίσουμε αύριο. Να ακυρώσουμε το ψήφισμα διότι βασίζεται σε περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όπως μας κατέδειξε η παρέμβαση της Επιτρόπου. Καλό λοιπόν το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή άτυπα να έρθουν σε επαφή με τη διάσκεψη των Προέδρων ώστε να γίνει η απαραίτητη ανταλλαγή απόψεων ώστε αύριο στην αίθουσα πριν από τα ψηφίσματα να ψηφίσουμε την, αψο... την απόφαση να μην ψηφίσουμε τα ψηφίσματα και να ε, περιορίσουμε τη συζήτηση μόνο σε ιδεολογικά στοιχεία. Thank you, Chairman. Madam... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να μιλήσω τώρα στα ρωμανικά. κυρία Επίτροπος, επιβεβαιώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε δίκιο που ε, ξεφράστηκε κατά του νόμου για τα ΜΜΕ στην Ουγγαρία. Το... Η Ουγγρική κυβέρνηση τώρα εξέφρασε την βούλησή της να τροποποιήσει τέσσερα ε, κεφάλαια του νόμου αυτού που είναι αντικείμενο αντιδημοκρατικής προσέγγισης. Αναλύθηκε η νομοθεσία αυτή και συμβατότητας με την κοινοτική νομοθεσία. Και θα ήθελα να μας πείτε ότι θα αναφερθείτε στην, ε, στον, στη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, Επιτροπή, πώς είναι δυνατόν να θεωρήσετε ότι πρότυπα της Ευρωπαϊκής Χάρτας ε, ξεπερνάνε τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός αυτού, εάν κάποια άλλη χώρα είχε ε, νέα νομοθεσία σύμφωνη με αυτή την αρχική νομοθεσία της ε, Ουγγαρίας θα αναγνωρίζετε ότι ήταν εσφάλμα της. Πάνω. Ο κύριος Σπάσκα, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ Μαρτώνη. Στη Σλοβακία έχουν ε, μια παροιμία που λέει ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι καλυμμένος με καλές προσθέσεις. Ε, δεν θέλω να διαφυσβητήσω την καλή πρόθεση των Ούγγρων φίλων μας, αλλά θα ήταν ίσως ευκταίο να είμαστε πιο προσεκτικοί όσον αφορά κάποιες διατυπώσεις. Πολλές από τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που προβλέπει η Ουγγαρία ο, μας κάνουν να ξεχνάμε κάποια πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για την διπλή υπηκότητα. Γιατί και εδώ θα υπάρξουν πολλά προβλήματα. Οι φίλοι μας στο Καναδά ή στην Αμερική, τι θα, ε, πώς θα αντιδρούσαν αν εκατοντάδες χιλιάδων Σέρβων ή Ουκρανών ερχόντουσαν στη χώρα τους όταν τους είχαν δώσει διαβατήρια για να πάνε μέχρι την Ουγγαρία. Δεν ξέρω, υπήρχε πραγματικά σκαλή πρόθεση. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μέσα στο νόμο αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι κατοχυρώνεται πλήρης κάλυψη των γεγονότων. Καλό φαίνεται αυτό. Επίση, προβλέπονται κυρώσει όταν παραβιάζεται το δημόσιο συμφέρον, αναταράσσει τη δημόσια τάξη. Είναι λίγο ασαφεί αυτέ οι ιδέε και άρα είναι επικίνδυνε. Εξίσου επικίνδυνε όπω και ο ρατσισμό και η ξενοφοβία. Μα κανεί όμω δεν νομοθετεί κατά αυτόν. Οπότε, γιατί λιθοβολούμε την Ουγγαρία και δεν κοιτάζουμε τα πρότυπα ε, σχετικά με την ελευθερία στι δικέ μα ε, χώρε. Ε, η BBC, παραδείγματο χάρη, κάνει ο μιλητής ένα λογοπαίγνιο για τα αρχικά, αμετάφραστο, και ε, ε, αντιμετωπίζει χειρότερα προβλήματα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα ανάλογα με ποιου ε, προσκαλούν ας πούμε, σε εκπομπέ και σε ποιου ε, δεν ε, προσκαλούν. Ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να κινητοποιηθούμε και στι δικέ μα τι χώρε. Η Επίτροπο, η κυρία Η Επίτροπος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κάποια μέλη έθεσαν την ερώτηση και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα κατά πόσον είναι σύμπτωση το σημερινό χρονοδιάγραμμα. Ήταν προσχεδιασμένο να επιληθεί το θέμα με την Ουγγρική κυβέρνηση σήμερα. Ορισμένες φορές χρειάζεται κάποιος ένα απαλό άγγιγμα στο νόμο και συμφωνώ κι εγώ Και εγώ θα προτιμούσα όταν με καλείτε να διευκρινίσω τι διακυβεύεται, να μπορώ να έρθω εδώ και να σας μιλήσω με απτά στοιχεία. Το κατά πόσον είναι σύμπτωση λοιπόν, κατά κάποιον τρόπο, και αυτό σας το λέω έτσι εν θερμό, μιλάμε για μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου και βρισκόμαστε πλέον στα μέσα Φεβρουαρίου. Περίπου 7 εβδομάδες διέρχησε, λίγο παραπάνω στα έξι χρόνια που βρίσκομαι ε, εγώ σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς νομίζω ότι ε, η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί έως και ταχεία. Από πείρα δεν ε, επιλύονται τόσο γρήγορα αυτά τα προβλήματα. Φοβούμαι ότι σπάνια μπορούμε να λύσουμε προβλήματα εντός επτά εβδομάδων. Πέραν αυτού όμως είναι και συναρπαστικό το να μάθουμε ποιο είναι το όλο υπόβαθρο, πώ προέκυψε η λύση. Πρόκειται για συνδυασμό κύριε Πρόεδρε, για συνδυασμό πραγμάτων και δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε το θέμα αυτό. Με έχετε προσκαλέσει εδώ και στο παρελθόν. Ήσασταν σαφεί, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το τι διακυβεύεται, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το τι ακριβώς ε, σκέφτεται κάθε πολιτική ομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και συζητάμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας εξηγήσω ότι το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του τύπου, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήταν, αν μη τι άλλο, γελίο ε, να μην το θεωρήσουμε βασική προτεραιότητα, να μην θεωρήσουμε βασική προτεραιότητα την προάσπιση της δημοκρατίας. Το κατά πόσον ήταν σύμπτωση το γεγονός ότι το προηγούμενο θέμα που είχατε εσείς στην ημερήσια διάταξη ήταν η Αίγυπτος και η δημιουργία μιας νέας δημοκρατίας. Νομίζω ότι μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα γνωρίζει όλα αυτά και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να προασπίσουμε και να επανορθώσουμε όπου ίσως υπάρχει επίθεση στη δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, το τρίτο θέμα είναι φυσικά η Ουγγρική Προεδρία. Ας μην είμαστε αφελείς. Σαφώς οι φίλοι ενός κράτους μέλους της οικογένειας της Ευρώπης γνωρίζουν ότι ε, το να είναι κάποιος στην Προεδρία είναι λίγο πολύ υποχρέωση. Από πλευράς τους λοιπόν υπήρχε μία ε, στάση ε, η οποία έλεγε ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Και μια τελευταία εξήγηση από πλευρά μου, αφού μου ζητάτε να δώσω εξηγήσει, είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν σαφέστατο. Ε, γράψατε, δώσατε πληροφορίες προς τον ε, υπόλοιπο κόσμο μέσω του τύπου, μέσω του ελεύθερου τύπου όπως είπατε κι εσείς. Επομένως μην υπατιμάτε το ρόλο σας. Πέραν αυτού όλο ο συνδυασμό αυτών των πραγμάτων εν τέλει για μένα αποτελεί και την εξήγηση γιατί βρισκόμαστε εδώ σήμερα με αυτό ε, το θέμα στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα τώρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και μην παρουσιάζετε επιχειρήματα ότι εγώ μόνο ενδιαφέρομαι για την ειρήνη και την ε, ηρεμία μάλλον δεν με ξέρετε καθόλου, διότι εγώ είμαι αυτή η οποία υπεραμείνεται της δημοκρατίας και έχω και κάποια πείρα επί του θέματος ε, ε, και μια μακρά ζωή ε, σε σχέση με τους περισσότερους από εσά στα θέματα της πολιτικής. Να σας αναφέρω τώρα κάποια θέματα τι γίνεται με την ανεξαρτησία του ρυθμιστή των ε, μέσων ενημέρωση. Η προκαταρκτική ανάλυση που κάναμε, κύριε Πρόεδρε, στην Ουγγρική νομοθεσία καθορίζει ότι ο τρόπος εκλογές και επιλογής ε, του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι αντίστοιχος με αυτούς οι ε, οποίοι είναι κοινά αποδεκτοί στην Ευρώπη. Έχουμε μία ε, πρόκληση πρέπει να αναγνωρίσουμε, ορισμένες φορές επαφιέται σε εσά, ορισμένες φορές όχι, ότι η Ουγγρική κυβέρνηση έχει μια πλειοψηφία δύο τρίτων και αυτό στη δημοκρατία είναι γεγονός. Η εφαρμογή του άρθρου 11. Εμείς εφαρμόζουμε την οδηγία, την οδηγία VMS και τη συνθήκη και Φυσικά συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο 11 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Δεν υπάρχει καμία δικαστική αναθεώρηση της απόφασης ε, του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, όπως έλεγε ο συνάδελφος Μωράες. Η απόφαση του Συμβουλίου των Μέσων είναι απόφαση πρωτόδικη και δεν μπορεί να ε, υπάρξει έφεση κατά της διαδικασίας αυτής αλλά όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 η επίσημη απόφαση του Συμβουλίου των Μέσων μπορεί να αμφισβητηθεί στο δικαστήριο βάσει των διατάξεων για τον κώδικα ποινικής ε, συγγνωμιαστική διαδικασίας και δεν θα πρέπει να υπάρχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, αλλά ε, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης απόφασης. Κύριε Βέμπερ, η προστασία των πηγών στον ε, νόμο της Ουγγαρίας είναι ανεπαρκής μας λέτε. Αν θεωρήσουμε την ελευθερία των μέσων ως βασική ευρωπαϊκή αρχή, όπως σας είπα στην αρχική μου παρέμβαση, αυτή θα πρέπει να είναι η αρχή αλλά και το τέλος όλου αυτού του ζητήματος και πάντα ήμουν υπέρ αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συνεχίσω να το υπερασπίζομαι. Σας το υπόσχομαι αυτό, θα συνεχίσουμε να προάγουμε συνεχώς το θέμα αυτό. Το δικαίωμα του δημοσιογράφου να προστατεύει τι πηγέ του σαφώ είναι μία από τι βασικέ αρχέ που διασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση τη ελευθερία του τύπου. Οι δημοσιογράφοι δεν θα πρέπει ποτέ να απαιτείται να αποκαλύπτουν τις πηγές τους εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για ποινική έρευνα. Και αυτή η αρχή Κύριε Πρόεδρε, είναι έγκυρη οποιοδήποτε και αν είναι το πολιτικό κλίμα που επικρατεί και μάλιστα θα, να πω, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να την υπερασπιζόμαστε με περισσότερο πάθος όταν ο τύπος και τα ΜΜΕ είναι σε πιο αδύναμη θέση όπως ισχύει σήμερα. Και όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη σχετική νομοθεσία, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών. Ωστόσο, η οδηγία δεν ισχύει σε δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των ευρωπαϊκών συνθήκων. Και αυτό είναι γεγονός. Και αυτό σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν ισχύει για θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την κρατική ασφάλεια και την επιβολή του ποινικού δικαίου. Και σύμφωνα με τις αρχές της ε, επικουρικότητας, τα κρατημέλη έχουν την ευθύνη να εξετάσουν ζητήματα που μπορεί να επηρεάζουν ε, την ιδιωτική ζωή του ατόμου με βάση τους δικούς τους κανόνες και τις διεθνείς ευρωπαϊκές, και ευρωπαϊκές συμβάσεις σε σχέση με τις ατομικές ελευθερίες. Κάθε ποινή θα πρέπει, κύρωση θα πρέπει να είναι αντίστοιχη και ανάλογη με μια δημοκρατική κοινωνία και η Επίτροπο, ο Επίτροπος δεν μπορεί να έχει αντίρρηση το να καταδικάζει εθνικές νομοθεσίες απουσία της αναφοράς στο άρθρο 30 που αρκετοί ρώτησαν, αρκετοί ευρωβουλευτές το ρώτησαν. Ξέρω πως πολύ λυπάστε που η Κομισιόν δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη το άρθρο 30 όταν εξετάζει την νομοθεσία περί μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όμω αυτό δεν ισχύει. Και θα ήθελα να πω ότι Είναι ξεκάθαρο για μας ότι απλώς δεν ισχύει. Ωστόσο, στην αρχική μας πρόταση για την οδηγία είχαμε συμπεριλάβει μια υποχρέωση για τα κρατημέλη ώστε να εγγυώνται την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Και εσείς, και έχετε πολύ καλή μνήμη, όπως διαπιστώνω πολύ συχνά, η διάταξη αυτή δεν υποστηρίχθηκε από το Σύμβουλιο και παρά την ε, στεναρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία γνωρίζω, άλλαξε στην σημερινή μορφή του άρθρου 30 της ε, οδηγίας τελευταία τύπωση δεν θεσπίζει υποχρέωση για τη δημιουργία ανεξαρτήτων σωμάτων. Κύριε Πρόεδρε, Δεν είναι αυτό που επιθυμούσαμε ακριβώ, αλλά αυτό είναι που υπάρχει σε αυτό το έγγραφο και εδώ θα πρέπει να δεχτούμε την πραγματικότητα, ακόμα και αν δεν μα ικανοποιεί απόλυτα. Οι Ουγγρικέ Αρχέ έχουν ε, διαγράψει την διάταξη στο εξή ε, αριθμιστικό ε, κείμενο του συντάγματος περί ΜΜΕ. Είναι υποχρέωση του συστήματος των ΜΜΕ να δίνει να παρέχει ακριβείς και αυθεντικές ε, αναφορές για τα γεγονότα. Αυτό λοιπόν θα ε, προσθεθεί μετά τις αλλαγές και θα ζητώ συγγνώμη που δεν είχατε το κείμενο, αλλά είχα και εγώ το κείμενο το οποίο διαπραγματευόμαστε, αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορούσα να σας το διαβιβάσω. Μόλις αυτό θα είναι δυνατόν. Θα σας το δώσω φυσικά, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς θα πιστέψετε τα όσα σας λέω και θα το εκτιμούσα αυτό ιδιαίτερος, αλλά και ότι τελικά θα το θέλατε και γραπτό, ώστε να έχετε την ευκαιρία να το διαβάσετε. Αυτό είναι ένα από αυτά τα ζητήματα που έχουν νόημα, ώστε και εσείς να αποφασίσετε. Δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση για ισόρροπη αντιστάθμιση στα γραπτά μέσα και στα οπτικοακουστικά. Και αυτό το είπα ήδη στις ε, αρχικές μου παρατηρήσεις. Η ερώτηση που έθεσε ο κύριος Λόκεκαρντ, κατά πόσο είμαι έτοιμη να, υποβα... να προτείνω νομοθεσία για τον πλουραλισμό των ΜΜΕ, το είπα στην αρτήριά μου εισήγηση ότι είμαι έτοιμη να προβώ σε δράση στο τομέα του πλουραλισμού των ΜΜΕ με όλες τις αρμοδιότητες που έχω στη διαθέσή μου. Δεν ε, ε, μπορούμε να έχουμε την ίδια προσέγγιση για όλους, αυτό είναι ξεκάθαρο και η, το, η γκρική υπόθεση το κατέστησε αυτό ακόμα πιο σαφές. Εγώ έχω δημιουργήσει μια ομάδα εργασία. σας ευχαριστώ για την προθυμία που δείξατε να μπείτε και εσείς σε αυτήν την ομάδα εργασία για να συζητήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει μια ε, ολοκληρωμένη εικόνα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να ενεργήσουμε και αντιστοίχως πράγμα που θα συμπεριλαμβάνει και την ανεξαρτησία των ΜΜΕ. Θα είναι μία από τις μεγάλες μας προτεραιότητες. Η θέση του ΟΣΕ για την Ουγγρική νομοθεσία περί ΜΜΕ και η ανάλυση τους είναι ότι υπάρχει νομική βάση. Υπάρχει μάλλον ε, διαφορετική νομική βάση από την ανάλυση εκείνη και αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους, κύριε Πρόεδρε και οι κύριοι λόγοι που αναφέρει η ΟΑΣΕ είναι η ανησυχία της νέας αρχής περί ΜΜΕ, δηλαδή η μακρά διάρκεια θητείας των μελών τους και το ρύθμιση της ε, υπηρεσίας εκπομπών και νομίζω ότι αυτό μπορεί να ισχύει και στα μέλη άλλων ε, διοικητικών συμβουλίων των ε, υπηρεσιών ε, των τηλεοπτικών μάλλον υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό που διακυβεύεται και αυτή είναι και η τελική μου παρατήρηση κύριε Πρόεδρε είναι ότι το μήνυμα του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης και είμαι βέβαιος ότι ο Υπουργός Εξωτερικών θα επαναλάβει το μήνυμα αυτό στην Ουγγρική κυβέρνηση. Είναι ποια είναι η ακριβή του θέση. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στις 7 εβδομάδες όπου στενά συνεργαστήκαμε, ότι εγώ εντυπωσιάστηκα από τη συμβολή Το επιτελείο μου που ανέκαθεν δουλεύει πολύ σκληρά, αλλά σε αυτή την περίπτωση εντυπωσιάστηκα και από τις δύο πλευρά, πλευρές, γιατί επικοδομητικά συνεργάστηκαν ώστε να βρεθεί μια λύση, διότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να βρεθεί λύση. Ευχαριστώ. τέλος, ε, εξ ονόματος του... What? have a point of ε, ε, Ο κύριος Μαύρο, πρόεδρε, εγώ θέλω να καλέσω την Επίτροπο για διαδικαστικό θέμα να μας δώσει απόψε τα κείμενα στα οποία αναφερόταν, τουλάχιστον στους πρόεδρους των ομάδων, ώστε τουλάχιστον αύριο να μπορέσουμε νυφάλια να τα μελετήσουμε πριν να χρειαστεί να ψηφίσουμε. Επίτροπε, έχετε απάντηση. Όσον αφορά την απάντησή μου είναι προφανώς όχι και αντιλαμβάνομαι ότι και ο Υπουργός συνενεί Οπότε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα θα σας έρθουν. Πέραν ε, της ε, συνενέσεως ε, και του νεύματος, ο Υπουργός Εξωτερικών εκπρόσωπος του Συμβουλίου θέλει να λάβει και το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιώ το σώμα μου ή τα νεύματά μου για να εκφράσω την άποψή μου. Οπότε εδώ ε, εν ονόματι της Ουγγαρίας θα μιλήσω παρακαλώ και θέλω να ε, κάνω ορισμένα σχόλια διότι η απάντηση της Επιτρόπου Κρούς ήταν ε, εκτενής και λεπτομερέστατη ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο για τα Μέσα Ενημέρωσης και αυτό απαντήθηκε εάν δεν απατώμε οπότε μπορώ να περιοριστώ σε λίγα μόνο θέματα. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι η Ουγγαρία είναι δεσμευμένη ε, να εφαρμόσει τις αξίες, τις αρχές και τους κανόνες οι οποίοι προβλέπονται στο χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε όλα τα άλλα μέσα διεθνούς δικαίου και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν παρουσιάστηκαν οι πρώτες αυστηρές κρίσεις σχετικά με το νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, και αυτό ήταν πριν από την ε, ε, υιοθέτηση της νομοθεσίας και εδώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στον εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ και εγώ το μόνο που επιθυμούσα ήταν να δω, να αναλύσω το κείμενο και στη συνέχεια να μας πει ο κύριος αυτό αμφιβολίες είχε σχετικά με το κείμενο ή σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Γι' αυτό και αμέσως ε, στηρίξαμε την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ο θεματοφύλακας των ε, συνθήκων για να μας πει αν είχε συγκεκριμένες ε, αμφιβολίες και ανησυχίες. Αυτό όντως έγινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά την νομοθεσία, διατύπωσε προτάσεις οι οποίες όλες υιοθετήθηκαν και μπορώ εδώ να επιβεβαιώσω ότι μεθαύριο θα συνέλθει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα εγκρίνουμε το κείμενο και θα υποβληθεί άμεσα προς ψήφιση από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και οι τροπολογίες θα υιοθετηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα από πλευράς διαδικασίας για να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σκληρή δουλειά της ε, για την ε, βοήθεια και στήριξή της και θέλω να ευχαριστήσω και όλους από εσά ε, διατύπωσαν λογικά σχόλια και μας βοήθησαν κατά αυτήν την διαδικασία η οποία είμαι βέβαιος ότι είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για τη χώρα μου αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Θα ήθελα λοιπόν απλώς να προσφέρω τη βοήθειά μου και την πλήρη στήριξή μας στην ομάδα αυτή εργασία στην οποία θα καταρτήσετε η κυρία Επίτροπε. Νομίζω ότι είναι προς όφελος όλης της Ευρώπης. Θέλουμε να συμμετάσχουμε και να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Το μόνο το οποίο λυπούμε είναι οι παρεκτροπές, οι λεκτικές παρεκτροπές που είδαμε σε ορισμένα Ευχαριστώ δηλώσεις ε, γιατί είχαμε ορισμένες φορές ε, την εντύπωση ότι μας ε, γίνεται αυτό που λέγουν οι, οι Γάλλοι προσέντεν των σιών δηλαδή μας είχαν προκαταλάβει ως ενόχους ενώ πρέπει ο καθένας να θεωρείται ως αθώος μέχρι ότου υποβληθεί σε μία δίκαιη η δίκη. Για το λόγο αυτό υπήρξε και η πολιτική συζήτηση, η οποία όμως πολιτική συζήτηση που όπως σας είπα στηρίζει στηρίχθηκε σε ε, ευρωπαϊκό και γενικό επίπεδο όντως ε, ίσως ε, ε, ήταν εις βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων και της ολοκλήρωσης της Ευρώπης αλλά τώρα αυτά είναι παρελθόν και θέλω και πάλι να επαναλάβω τον σεβασμό τον οποίο έχουμε και να σας πω ότι σκοπεύουμε να ενσωματώσουμε το χάρτη των ουσιαστικών δικαιωμάτων στον στο νέο σύνταγμα της Ουγγαρίας διότι είναι η πρώτη χώρα όπου ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα αποτελέσει ε, μέρος ε, του ε, του συνταγματός και ε, θα προέχει ιεραρχικά από οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία ε, όποια και να είναι αυτή, ε, από οποιοδήποτε θέματος και ε, πιστεύω ότι αυτό θα βεβαιώσει όλους σας ότι οι θεμελιώδεις ε, αξίες και οι θεμελιώδεις αρχές τις οποίες συμμεριζόμαστε όλοι ε, θα εφαρμοστούν και θα γίνουν σεβαστές στη χώρα μου. Σας ευχαριστώ. Έλαβε έξι προτάσεις ψηφίσματος για την περνάτωση της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε αγαπητοί συνάδελφοι. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα ενός λεπτού για να έρθει ο επόμενος αρμόδιος ο και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το επόμενο θέμα που αφορά στην Κορέα.